Uh, Συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, ας ξεκινήσουμε παρακαλώ. Καθίστε αν θέλετε. Well, let's open. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε. Ξεκινά το δεύτερο τμήμα της συνεδρίασης μας που ξεκίνησε χτες. Και περνάμε στο 13 σχέσεις, οικονομικές και εμπορικές σχέσεις ΕΕ Μεξικού. Ας ξεκινήσω καλωσορίζοντα πρώτα την εξοχότητά του τον πρέσβη του Μεξικού στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τον κύριο Χουάν Χωσέ Γκόμες, που πρόσφατα διορίστηκε ως πρέσβης. Είχαμε ήδη το προνόμιο να συναντηθούμε πρόσφατα μαζί του και αποδέχθηκε την πρόσκλησή μας να προσέλθει εδώ για μια ανταλλαγή απόψεων για τα θέματα των οικονομικών και εμπορικών σχέσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης και Μεξικού. Το Μεξικό, όπως θα θυμόσαστε, θα ήθελα να σας υπενθυμίσω, έχει εκφράσει το ενδιαφέρον του να εξυγχρονίσει την συμφωνία πλαίσιο για το εμπόριο, σφαιρική συμφωνία, Global Agreement, με διατάξεις που ε, είχαν εκπονηθεί που για μια συμφωνία που άρχισε να ισχύει τον Οκτώβριο 2000 για τα τμήματα που αφορούν το εμπόριο σε σχέση με τα αγαθά και στη συνέχεια για τις υπηρεσίες όσον αφορά τον εξυγχρονισμό αυτής της συμφωνίας αρκετές συνεδριάσεις έχουν λάβει χώρα σε τεχνικό επίπεδο ήδη για να αξιολογηθεί, να σταθμιστούν οι δυνατότητες του εξυγχρονισμού αυτής της συμφωνίας. Μετά την συνεδρίαση της Επιτροπής Εμπορίου τον Ιούνιο πέρυσι υπάρχει πολιτική βούληση να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα και η κατάσταση συνολικά για να μπορέσει να εξυγχρονιστεί το πλαίσιο αυτό, το νομικό πλαίσιο των εμπορικών μας σχέσεων με το Μεξικό. Φυσικά πρέπει να είναι σαφές ότι ο εξυγχρονισμός θα προσφέρει πρόσθετη αξία σε σχέση με την ενισχύ σημερινή κατάσταση ως έχει. Και η ομάδα εποπτείας σε σχέση με το Μεξικό παρακολουθούσε, παρακολούθησε αυτές τις συζητήσεις η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου ενέκρινε μια προφορική ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή από αυτού του θέματος που εγκρίθηκε από το Κοινοβούλιο τον Ιανουάριο εφέτος. Έτσι το Κοινοβούλιο εξέφρασε μια θετική τοποθέτηση και άποψη σε σχέση με τον εξυγχρονισμό, την επικαιροποίηση καλύτερα αυτής της συμφωνίας υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι το επίπεδο φιλοδοξιών πρέπει να αντιστοιχεί στη νέα γενεά εμπορικών συμφωνιών που συνάπτει και συνήψε η Ευρωπαϊκή Ένωση με άλλες χώρες. Για παράδειγμα τα τελευταία χρόνια με την Νότια Κορέα, Περού, Κολομβία και τα λοιπά. Επιτρέψτε μου τώρα να δώσω τον λόγο στον πρέσβη του Μεξικού, τον κύριο Γκόμες. Κύριε πρέσβη, καλώς ήρθατε, σας ευχαριστούμε που ήρθατε, έχετε τον λόγο. Παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, καλή σας μέρα. Αξιότιμα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου. Σε σχέση με εξ του Μεξικού, εκτιμώ ιδιαίτερα, εκφράζω την ιδιαίτερη εκτίμηση μου προς εμάς κύριε Πρόεδρε, που είχα τη μεγάλη τιμή να συναντηθώ μαζί σας πρόσφατα και το μου στείλατε αυτή την πρόσκληση για να μπορέσω να συζητήσω κάπως μαζί σας για το πού βρισκόμαστε, πού βρίσκεται σήμερα το Μεξικό σε αυτό το πλαίσιο. Επιτρέψτε μου να επικαιροποιήσω κάποια στιγμιότυπα, κάποιες εικόνες για παράδειγμα σε σχέση με το πλαίσιο αυτής της διαδικασίας επικαιροποίηση αυτής της συμφωνίας που εσείς πολύ καλά αναφέρατε προηγούμενα. Η κυβέρνηση του Μεξικού, Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη, δέχτηκε με ιδιαίτερη ευχαρίστηση την πρόταση των κυρίων Προέδρων Φαν Ρόμπαϊ και Μπαρόζο ώστε ακριβώς να ξεκινήσει η διαδικασία επικαιροποίηση της σφαιρικής ε, ολοκληρωμένης συμφωνίας, ιδιαίτερα της εμπορικής συμφωνίας. Και ο λόγος για τον οποίο η κυβέρνηση του Μεξικού και ο πρόεδρος άμεσα δέχτηκαν αυτή την πρόταση, συσχετίζεται μεταξύ άλλων λόγων με το ότι το Μεξικό κατά τα τελευταία 15-20 χρόνια εισήλθε σε μια διαδικασία σε βάθος μεταρρύθμισης οικονομικής και πολιτικής που είναι φυσικό ότι δημιούργησε και το ίδιο συμβαίνει και σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση το όχημα που είχαμε μεταξύ των δύο μελών για το εμπόριο και εσείς το αναφέρατε είναι λιγότερο πλέον αποτελεσματικό η παλαιά συμφωνία για να υποφεληθούμε όσον αφορά τις νέες ε, νεότερες ευκαιρίες. Λοιπόν Πρόεδρε απλά και μόνο θα ήθελα να κάνω μια περιγραφή εν συντομία του πού βρίσκεται σήμερα το Μεξικό και να ολοκληρώσω ίσως με κάποια σχόλια, κάποιες παρατηρήσεις σε σχέση με τις αυστηρότερα θα έλεγα εμπορικές πτυχές. Όπως γνωρίζετε και είσαστε πολύ καλός γνώστης της χώρας μου, κυρίως από τα τέλη της δεκαετίας του 80 και τη δεκαετία του 90 ξεκίνησε το Μεξικό μία από τις φάσεις μεταμόρφωσης, μεταρρύθμισης οικονομικής, πιο, μία από τις πιο έντονες στην ιστορία του Μεξικού, όπου επιτυγχάνεται κυρίως ξεκινά η οικοδόμηση ενός συστήματος, μιας πολιτικής και ενός οράματος για τα δημοσία οικονομικά και τα νομισματικά θέματα γενικότερα και το μακροοικονομικό σύστημα που <clears throat> με την πάροδο των ετών διασφάλισε ότι σήμερα το Μεξικό έχει και εδώ και το διάστημα ένα μακροοικονομικό σύστημα στη διάθεσή του ε, ιδιαίτερα ενδυναμωμένο, είναι ιδιαίτερα αναζωογονημένο. Έχουμε πολύ υγιή δημοσιονομικά και στο νομισματικό και στο δημοσιονομικό τομέα. Κάποιες σημαντικές ίσως παρατηρήσεις για αυτό το θέμα θα ήταν ότι στα δημόσια οικονομικά και στα μακροοικονομικά θέματα εδώ και αρκετά πολλά χρόνια στο Μεξικό έπαψαν να υπάρχουν πολιτικές συζητήσεις γύρω από αυτά. Εδώ και πολλά χρόνια στο Μεξικό οι πολιτικές δυνάμεις της χώρας μου δέχονται ότι η ενδυνάμωση των δημοσίων οικονομικών, η, η εξυγίανση, η μακροοικονομική και δημοσιονομική είναι απλά και αποδεκτή ως μια πολιτική, κρατική πολιτική που πρέπει να προαχθεί. Άσχετα από το πολιτικό προφίλ και τις ιδεολογικές τοποθετήσεις των κομμάτων στην Βουλή του Μεξικού, η συζήτηση που διεξάγεται είναι ένα θέμα αυτονόητο αυτό, το οποίο αποδέχονται όλοι. Και αυτό μας επέτρεψε σίγουρα <clears throat> να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε τις ε, πρόσφατες οικονομικές κρίσεις, θα έλεγα με έναν πάγιο και υγιή τρόπο και με μεγάλη νυφαλιότητα και το 2009 σημειώθηκε μια δραματική πτώση αρκετών ποσοστιών μονάδων ε, στο Μεξικό και ταυτόχρονα υπήρξε μια δραματική ανάκαμψη θα έλεγα ξεχωριστή ανάκαμψη λόγω της ε, ε, ενδυναμωμένης δημοσιονομικής κατάστασης ισχυρής δημοσιονομικής κατάστασης σε σχέση λοιπόν με το Κοινοβούλιο και την, και την Επιτροπή είναι η οικονομική ανάπτυξη η πρόοδος και από πλευράς των δυνάμεων πολιτικών και της ε, κυβέρνησης αυτή η ανάπτυξη, η οικονομική ανάπτυξη περνά ακριβώς από την παραγωγικότητα, την αύξηση της παραγωγικότητας, την ανταγωνιστικότητα, την αύξηση της ανταγωνιστικότητας και την καινοτομία. Και για να πετύχουμε την καινοτομία, την ανταγωνιστικότητα και την παραγωγικότητα στο Μεξικό που θα εγγυώνται μια υφόρο ανάπτυξη μακροπρόθεσμα, χρειαζόμαστε, έπρεπε να περάσουμε σε μια διαδικασία σε βάθος, έντονη διαδικασία εξυγχρονισμού θεσμικού και δομικών διαθροτικών αλλαγών, μεταρρυθμίσεων. Εύκολα λέγεται κάτι τέτοιο, αλλά γνωρίζετε ότι κάτι τέτοιο είναι ιδιαίτερα περίπλοκο σε μια χώρα που έχει επιπλέον και τα χαρακτηριστικά του Μεξικού. Μια πολύ μεγάλη χώρα με 120 εκατομμύρια κατοίκους, που είμαστε μία από τις οικονομίες, μία από τις μεγαλύτερες οικονομίες παγκόσμια και εξάγουμε, είμαστε από τους μεγαλύτερους ε, εξαγωγείς και εισαγωγείς ταυτόχρονα παγκόσμια, από τους μεγαλύτερους. Έτσι λοιπόν όταν ξεκίνησε η κυβέρνηση του κυρίου Πρόεδρου Πένια ο Πρόεδρος ε, ηγήθηκε αυτής της ε, διάρθρωσης της πολιτικής υπέρ του Μεξικού που είναι όπως την αποκαλούμε ένα εγχείρημα που συνενώνει όλες τις δυνάμεις στο Κογκρέσο του Μεξικού όλων των πολιτικών δυνάμεων και μέσω του οποίου αυτού εγχειρήματο <clears throat> δόθηκε η έγκριση σε σχέση με το εγχείρημα του Προέδρου συμφωνήθηκαν ε, οι στόχοι που θα έπρεπε να υλοποιηθούν για να μπορέσει το Μεξικό να κάνει αυτό το άλμα, να ενδυναμώσει τα δημοσιονομικά του και τα οικονομικά του ώστε να καταλήξει σε μια αηφόρο ανάπτυξη με την παραγωγικότητα, την ανταγωνιστικότητα που θα έπρεπε να ενισχυθούν και για όλα αυτά έπρεπε να εκπονηθεί ένα πρόγραμμα με ένα μεγάλο σύμφωνο που θα μπορούσε εγκάρσια να ε, ενώνει και να περνά από όλους τους τομείς για τον εξυγχρονισμό. Και με αυτόν τον τρόπο οι πολιτικές δυνάμεις συμφώνησαν σε πέντε μεγάλους στόχους που θα έπρεπε να επιτευχθούν. Ο πρώτος από αυτούς τους στόχους είναι ένα ειρηνικό Μεξικό, μια ειρηνική διαβίωση στο Μεξικό. Όλοι οι Μεξικανοί και όλες οι δραστηριότητες κοινωνικές και οικονομικές στη χώρα μας να μπορούν να αναπτυχθούν απόλυτα υπό το πλαίσιο του νόμου του κράτους δικαίου οπωσδήποτε. Και ο δεύτερος μεγάλος στόχος είναι όλοι οι Μεξικανοί πολίτες να μπορούμε και να πρέπει να έχουμε και τα παιδιά μας πρόσβαση και προσπελασιμότητα όχι μόνο σε μια ολοκληρωμένη σφαιρική παιδεία και εκπαίδευση που ήδη έχουν αυτήν την πρόσβαση αλλά κυρίως και αυτό είναι το πιο σημαντικό, μια παιδεία και εκπαίδευση ανώτατης ποιότητας, αναβαθμισμένη. Τρίτο, δεν μπορούμε να έχουμε το στόχο να πετύχουμε μια χώρα πιο εξυγχρονισμένη αν δεν έχουμε μια κοινωνία η οποία να εντάσσει στους κόλπους της όλους τους πολίτες της. Δεν μπορούν να υπάρχουν αποκλεισμοί, δεν μπορεί να υπάρχουν διαφορετικά ε, στρώματα και διαφορετικές κατηγορίες Μεξικανών. Όλοι οι Μεξικανοί πρέπει με ισοδύναμο, ίσο τρόπο να έχουν πρόσβαση σε όλα τα ωφέλη και τα προτερήματα τα οποία θα τους, θα τους προσφέρονται κοινωνικά και να μπορούν έτσι να συνεισφέρουν μέσα από ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο στην ανάπτυξη. Και επόμενο Τέταρτο, όπως προανέφερα, δεν μπορούμε να πετύχουμε τίποτα για όλα αυτά αν δεν δημιουργήσουμε ένα Μεξικό που να ευημερεί, ένα Μεξικό που να μπορεί να παράγει πλούτο, που να μπορεί να κατανέμεται με δίκαιο, ισοδίκαιο τρόπο μεταξύ όλων των κατοίκων του, μεταξύ των 120 εκατομμυρίων πολιτών. Και σίγουρα όχι μόνο είμαστε 120 εκατομμύρια πολίτες στο Μεξικό, αλλά η μέση ηλικία στο Μεξικό είναι 26 ετών των πολιτών μας. Έχουμε μια πολύ νέα λοιπόν όσον αφορά ηλικιακά την κοινωνία μας και μια προοπτική συνεισφοράς πολύ ενδυναμωμένη, τεράστια για την ανάπτυξη του Μεξικού και κυρίως με μεγάλες φιλοδοξίες. Και τέλος, ο πέμπτος στόχος που θέτει η Συμφωνία για το Μεξικό ενώπιον της είναι λόγω των διαστάσεων του Μεξικού και των ικανοτήτων του Μεξικού ως χώρας όπου το θεσμικό δυναμικό που έχουμε, η παρουσία μας σε παγκόσμιο επίπεδο, συνεπάγεται ότι πρέπει να δεχτούμε ότι θα πρέπει ανάλογα με αυτές τις διαστάσεις να επομισθούμε τις ευθύνες ε, υπεύθυνα σε ένα επίπεδο δηλαδή συνεισφοράς για την ανάπτυξη που συνεπάγεται δέσμευση, ένα αίσθημα υπευθυνότητας και ένα καθήκον συνολικό, πράγμα το οποίο θα δημιουργήσει τη δυνατότητα να συμμετάσχει το Μεξικό με αυτή την ιδέα της υπευθυνότητας και της ευθύνης, να συμμετέχει στην αντιμετώπιση των παγκόσμιων προκλήσεων. Ίσως ο καλύτερος τρόπος να το περιέγραφω αυτό θα ήταν ε, ότι εμείς ε, το κατανοούμε απόλυτα ότι η ευημερία του Μεξικού εξαρτάται από την ευημερία των υπόλοιπων. Δεν μπορεί να δημιουργηθεί ευημερία εν κενό και μπορεί η ευημερία να δεν μπορεί να υπάρξει ευημερία απομονωμένα ως νησίδα. Σε αυτόν τον παγκοσμιοποιημένο, αλληλεξατοποιημένο κόσμο η ευημερία του ενός πρέπει να είναι η ευημερία του άλλου. Και μέσα σε αυτό το συνολικό θέμα είναι ένα θέμα που έχει κέρια ε, σημασία για την κοινοβουλευτική σας επιτροπή. Διότι το εμπόριο ακριβώς και η ανάπτυξη και η ευημερία αποτελούν συλλογικούς στόχους ε, και φιλοδοξίες. Για να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι, Πρόεδρε, το Σύμφωνο για το Μεξικό, Πάκτο Πορμέχικο, συμφώνησε σε ένα πολύ εντυπωσιακό και πολύ φιλόδοξο πακέτο, δέσμης μέτρων δηλαδή, διαρθρωτικών ε, αλλαγών, που δεν είναι μόνο δεν είναι μόνο δομικές, αλλά είναι χαρακτήρα που θα μεταμορφώσουν το Μεξικό σε μια άλλη χώρα. Έτσι λοιπόν σε ένα ε, εδώ και ε, ένα μήνα ενέκρινε το, Συμβου... το... η Βουλή ένα πρόγραμμα μεταρρύθμισης ε, στα εργασιακά θέματα, στην εκπαίδευση και την παιδεία, μια μεταρρύθμιση και αλλαγές στα τηλεπικοινωνιακά, στα δημοσιονομικά επίσης άλλη μεταρρύθμιση, οικονομική μεταρρύθμιση επιπλέον, ένα πακέτο μέτρων όσον αφορά την ανταγωνιστικότητα στο οικονομικό επίπεδο, πολιτική εκλογική μεταρρύθμιση και ενεργειακή ή μεταρρύθμιση επίσης. Τις επόμενες λοιπόν εβδομάδες ε, θα υποβληθούν στο ε, Κογκρέσο του Μεξικού οι προτάσεις ε, για μια μεταρρύθμιση στον τομέα της αγροκτηνοτροφίας. Με αυτή την ομάδα κατηγορία ολόκληρη μεταρρυθμίσεων, όπως μπορείτε να δείτε, είναι μεταρρυθμίσεις πρώτων που εγκάρσια περνάνε σε όλη την ζωή οικονομική και κοινωνική του Μεξικού και την αφορούν άμεσα και αρθρώνονται και συνδυάζονται η μία μεταρρύθμιση με την άλλη, ώστε η μία να ενισχύει και να ενδυναμώνει την επόμενη, ώστε όλες αυτές στο τέλος συνολικά να μπορούν να αρθρώνονται σε ένα συνολικό ε, ολοκληρωμένο πλαίσιο και να ενισχύουν με εκθετικό τρόπο πολλαπλασιαστικά την ικανότητα του Μεξικού να παράξει αυτό το οποίο αναφέρθηκε στην αρχή. Μια οικονομική ανάπτυξη που θα βασίζεται στην καινοτομία, στην ανταγωνιστικότητα και στην παραγωγικότητα. Κύριε Πρόεδρε, το Μεξικό σήμερα εξάγει το 60% όλων των μεταποιημένων εξαγωγών του συνόλου της Λατινικής Αμερικής. Είναι μεγαλύτερο, μεγαλύτερος ο εμπορικός όγκος των εμπορικών σχέσεων και των εξαγωγών του Μεξικού από ό,τι της Νότιας Αμερικής. Ένα δισεκατομμύριο ε, δολάρια αγαθά εξάγουμε καθημερινά και πάνω από 80% αυτών των εξαγωγών είναι εξαγωγές μεταποιημένων προϊόντων που έχουν παραχθεί στο Μεξικό. Το η οικονομική λοιπόν ανάπτυξη του Μεξικού και η ανάπτυξη της ικανότητας αγοραστικής δύναμης της χώρας μας που είναι μια χώρα μέσου εισοδήματος κατηγορίας μέσου εισοδήματος και έχει φτάσει ανακεφαλή περίπου στα 17-18 χιλιάδες ε, ανα ε, άτομο, αναπολίτη και είμαστε μια αναπτυσσόμενη χώρα αλλά στο ανώτερο, ε, στην ανώτερη κατηγορία όσον αφορά το εισόδημά μας. Ο ένατος εισαγωγέας σε παγκόσμιο επίπεδο και όδος εξαγωγός σε παγκόσμιο επίπεδο. Είμαστε λοιπόν η δεύτερη εισαγωγή, εξαγωγής όσον αφορά τις ΕΠΑ. Είμαστε το τέταρτο εξαγωγό κράτος όσον αφορά τα οχήματα, τις εξαγωγές οχημάτων και το ίδιο ισχύει και για τις ε, τηλεοπτικές ε, συσκευές τηλεοράσεις. Είμαστε ο πρώτος στόχος ε, επενδύσεων, αλλοδαπών επενδύσεων παγκόσμια όσον αφορά τον τομέα της αεροδιαστημικής, όπου περίπου 300 επιχειρήσεις συνεισφέρουν επενδύοντας πολύ μεγάλα κεφάλαια στο Μεξικό. Σημειώνεται αύξηση 30% κατά τα τελευταία 5 χρόνια στο Μεξικό σε σχέση με αυτές τις επενδύσεις και αυτό ανταποκρίνεται στο δυναμικό που υπάρχει καινοτομία τεχνολογικής που ήδη υφίσταται στο Μεξικό και τους πόρους που παράγονται ε, και τα προϊόντα που είναι αναβαθμισμένα ανώτατης ποιότητας ε, και έχουμε και έναν τεράστιο αριθμό μηχανικών μηχανολόγων 120.000 μηχανολόγοι μηχανικοί ε, παίρνουν τα πτυχία τους από τα πανεπιστήμια μας και θα ήθελα να πω σε αυτή την την ε, οικονομική ανάπτυξη του ε, Μεξικού μεγαλώνει η πίτα που μπορεί να μοιραστεί. Και σε αυτή την ανάπτυξη αυτής της πίτας που μπορεί να μοιραστεί και να αναδιανεμηθεί, κυρίως όσον αφορά τις εισαγωγές, σε σχέση με το ότι μπορεί να ε, πολιθεί σε εμάς και πρέπει να είναι και συνεπές με μια διαδικασία πολυμορφοποίησης των εμπορικών μας σχέσεων που σε, στη μεγάλη του πλειοψηφία εξακολουθούν αυτές οι σχέσεις να αφορούν τις ΗΠΑ. Αλλά όλο και περισσότερο έχουμε και σχέσεις και με άλλες περιφερειέ και περιοχές και αγοράζουμε και αγαθά από τέτοιε τέτοιες περιοχέ περιοχές και περιφέρειες. Η πολυμορφοποίηση λοιπόν σε αυτό το τομέα υπήρξε με ραγδαίες εξελίξεις σημειώθηκε και θα ήθελα να πω σε αυτή την πολυμορφοποίηση κυρίως των εισαγωγών στο Μεξικό, αυτοί είναι οι χώροι που δημιουργούνται για πωλήσει προς το Μεξικό καταλήφθηκαν από χώρες της Ασίας στη συντηρητική τους πλειοψηφία. Η Ευρώπη δεν αύξησε τις εξαγωγές της ε, στο Μεξικό. Η Ευρώπη δεν επωφελήθηκε όπως θα έπρεπε αν επιθυμείτε, αν ε, θέλετε με αυτή τη ε, διατύπωση από την αύξηση της πίτας του Μεξικού. Ήταν η Κίνα, η Ιαπωνία, η Κορέα που επωφελήθηκαν. Ήταν οι χώρες της Ασίας που επωφελήθηκαν γενικότερα. Και όλα αυτά τι κάνουν καθιστούν όλο και περισσότερο προφανές ότι ο εξυγχρονισμός, η επικαιροποίηση της εμπορικής μας συμφωνίας έχει κάθε νόημα να γίνει και είναι πολύ σκόπιμο εγχείρημα. Και όπως σε ε, ξεχωριστούς φίλους και εταίρους στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και διμερός έχουμε πει, το Μεξικό δέχεται τις, προ... προτάσεις του των Προέδρων Φαν και Μπαρόζο. Και γι' αυτό εργαζόμαστε ακριβώς ε, και είμαστε πρόθυμοι να προωθήσουμε αυτό το θέμα με το μεγαλύτερο ενδιαφέρον, ώστε να συνεχιστεί και από την Επιτροπή με τον ίδιο τρόπο. Εκτιμώ ιδιαίτερα που μου δώσατε αυτή την ευκαιρία να σας προσφωνήσω, Πρόεδρε. Είμαι στη διάθεσή σας, αν χρειαστεί, για να απαντήσω σε σχόλια ή ερωτήσεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Πρέσβη για την παρουσίασή σας. Το έγγραφο αυτό έχει διανεμηθεί για τις διαφορετικές μεταρρυθμίσεις του Μεξικού και περιλαμβάνει τα όσα ανέφερε μόλις ε, ο προσκεκλημένος μας για την ενέργεια και τη τηλεπικοινωνία μεταξύ άλλων. Να δώσουμε τώρα το λόγο στα μέλη της ε, μόνιμης Επιτροπής ε, Παρακολούθησης για το Μεξικό. Βεβαίως έχουμε τον νόμιμο εισηγητή, τον κύριο από τους Σοσιαλιστές. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα, κύριε Πρέσβη, σα ε, καλωσορίζουμε στην Επιτροπή μας. Νομίζω ότι η εισήγησή σα δείχνει ότι το Μεξικό είναι έτοιμο να εισέλθει σε αυτές τις διαπραγματεύσεις. Όπως γνωρίζετε, ήμουν υπέρμαχο ε, αυτή τη συμφωνία και τη ε, αναβάθμιση τη. Γι' αυτό χαίρομαι που πηγαίνουν καλά οι συζητήσεις και η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Μεξικό αποφάσισαν την προηγούμενη εβδομάδα να εισέλθουν σε μια ε, τέτοια διερευνητική μελέτη και να εκπονηθεί και μία κοινή έκθεση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ξεκινήσει την ε, ε, αξιολόγηση των πυλώνων αυτών ως τμήμα της αξιολόγησης και ελπίζω στις αρχές του 2015 να έχουμε τα πρώτα αποτελέσματα. Πολλοί συνάδελφοι φαντάζομαι θα θέσουν ερωτήματα. Εγώ θα ήθελα μόνο να επικεντρωθώ σε δύο που είναι σημαντικά για την ομάδα μου. Πρώτον, για το κεφάλαιο αϊφόρος ανάπτυξη, που είναι σημαντικό, θεμελιώδους σημασία στοιχείο των εμπορικών συμφωνιών σήμερα και θα ήθελα να σας ρωτήσω εάν το Μεξικό είναι διατεθειμένο να διαπραγματευτεί την συμπερίληψη της βιώσιμης ανάπτυξης αυτού του κεφαλαίου, συμπεριλαμβανομένη στις Ρητρε των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, με έναν πλήρη ε, μηχανισμό για την εφαρμογή τη. Και το δεύτερο ερώτημα αφορά το μηχανισμό ε, ISDS, της επίλυση διαφορών. Γνωρίζετε ότι σήμερα βρισκόμαστε σε διαπραγματεύσεις με τις ΕΠΑ με το όνομα TTIP. Είναι ένα μεγάλο θέμα συζήτηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και για το κατά πόσο θα πρέπει να συμπεριληφθεί ο μηχανισμός ISDS. Θα ήθελα να μας πείτε ποια είναι η θέση του Μεξικού ε, για αυτό το θέμα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Από το ΕΛΚ. Ευχαριστώ Πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω για την παρουσία ανάμεσά μας του κύριου Πρέσβεως εδώ. Καλώς ήρθατε στην Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Σας ευχόμαστε κάθε επιτυχία σε αυτό το εγχείρημά σας, στην σταδιοδρομία σας. Θα ήθελα να τονίσω για άλλη μια φορά ότι πέρασε ένα έτος από την Σύνοδο Κορυφής του Αγίου Ιακώβου της Χιλής, όπου είχαμε την δέσμευση επικαιροποίηση τότε που αναλήφθηκε για την επικαιροποίηση συμφωνίας, ε, εμπορικής συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης Μεξικού. Πρέπει να πω ότι ικανοποιούμε, λέγοντας ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, ξεκίνησε μια μελέτη αξιολόγησης ε, για τις δυνατότητες αυτής της συμφωνίας και το ότι συμφωνήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα να ξεκινήσει αυτό το εγχείρημα το διερευνητικό στο Κοινοβούλιο έγιναν διάφορες ε, επαφές και τον προηγούμενο Ιανουάριο στην σύνοδό μας στο Στρασβούργο δεν είναι απόλυτα σαφές ποια δυνατότητα θα χρησιμοποιηθεί σε σχέση με τη ρήτρα αναθεώρησης ε, αυτή της συμφωνίας. Ίσως ο κύριος Πρέσβης θα μπορούσε να μας πει δύο λόγια για αυτό το θέμα. Και τώρα θα ήθελα να διατυπώσω δύο πιο εξειδικευμένε ερωτήσεις. Η μία η οποία αφορά την προστασία των επενδύσεων. Όπως γνωρίζετε <clears throat> κύριε Πρέσβη, αμφότερες οι πλευρές συμφωνούν ότι η συμφωνία αυτή πρέπει να διασφαλίζει έναν υψηλό βαθμό προστασίας των επενδύσεων συμπεριλαμβανομένου και ενός μηχανισμού επίλυσης ε, τριβών ε, και προβλημάτων ερώτηση ποια είναι η θέση του Μεξικού σε σχέση με αυτό το θέμα. Θα ήταν πρόθυμο να συμπεριλάβει τέτοιου είδου μηχανισμούς ε, ώστε να διασφαλιστεί η αύξηση της διαφάνειας ε, και της λογοδοσίας. Και ένα τελευταίο ερώτημα το οποίο συσχετίζεται με το θέμα το ενεργειακό. Γνωρίζουμε επίσης ότι αμφότερες οι πλευρές εξέφρασαν το ότι θα ήταν σπουδαίο, θα ήταν σημαντικό να συμπεριληφθεί σε αυτή τη νέα ε, συμφωνία να ενταχθούν θέματα τα οποία θα αφορούν τα ενεργειακά. Θα ήθελα να γνωρίζω ρωτήσω τι είδου μέτρα έχετε υπόψη για να γίνει κάτι τέτοιο. Ευχαριστώ. Thank you. Next. Ευχαριστούμε. Από την άλλη δεν βλέπω σκιώδη. Η άρη κύριε Μακλάρκιν. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, ευχαριστώ και τον κύριο Πρεσβευτή. Ε, άλλαξα θέση για να είμαι πιο κοντά, να σας βλέπω από κοντά. με τα χαράς ακούω το επίπεδο φιλοδοξιών ε, των σχεδίων σας και την πρόοδο που έχετε επιτύχει. Έχετε πραγματικά ε, πολλές δυνατότητες για το μέλλον. Είχα ε, συναντήσει και την κυρία Φουέντες στο παρελθόν, την προηγούμενη πρέσβη, και είχαμε συζητήσει τις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης και Μεξικού και η πολιτική θέληση ε, υποστήριζε πραγματικά ε, την ενίσχυση της ε, σχέσης του Μεξικού με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ισχύει αυτό πράγματι, υπάρχει αυτή η στήριξη. Συνεχίζεται αυτή η συζήτηση με τις πραγματεύσεις TTIP με τις ΕΠΑ. Ξέρουμε ότι και το Μεξικό θέλει να συμμετάσχει. Στις αρχές της εβδομάδας, εδώ πέρα στη συνεδρίαση, στο Κοινοβούλιο, με τον επικεφαλής των διαπραγματεύσεων, είχαμε δει τα θέματα που συζητούνται ε, και που εξετάζονται ξεχωριστά από κάθε τέρο. Εσείς ε, θα θέλατε να ε, διαμορφωθεί μία βορειοατλαντική εμπορική ομάδα, ας πούμε. Ευχαριστώ, ο κύριος Σόλτς. Από την ΚΟΕ, ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τον ε, κύριο Πρέσβη που μας ενημέρωσε για την ε, τρέχουσα κατάσταση και την ε, προετοιμασία του εδάφους σε ό,τι αφορά τις εμπορικές πραγματεύσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης και Μεξικού. 20 χρόνια μετά την ναύτα και πάνω από 10 χρόνια μετά την ε, Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, Μεξικού ήρθε η ώρα να εξετάσουμε πού βρισκόμαστε, ποιος ε, ήταν ο αντίκτυπος και ποια διδάγματα μπορούμε να αντλήσουμε από αυτή τη δεκαετή ολοκληρωμένη οικονομική συνεργασία και ποια ήταν τα ωφέλη για τους πολίτες και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού. Χθες είχαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα σε βάθος συζήτηση για το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ε, στις εμπορικέ ε, συμφωνίες και επενδυτικέ συμφωνίες με συμμετοχή ε, ακαδημαϊκού από το Πανεπιστήμιο του Cambridge. Ήταν μάλλον εντυπωσιακό το ότι υπάρχει σαφές αίτημα να συμπεριλαμβάνουμε δεσμεύσεις για την τήρηση της ρήτρας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις διεθνείς εμπορικές συμφωνίες. Βεβαίως, γνωρίζουμε τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η μεξικανική οικονομία, βεβαίως και οι οικονομίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης εν καιρό κρίσης. Πρέπει να αποφύγουμε παρόλα αυτά το κοινωνικό dumping, αλλά και την ε, καταπάτηση ανθρωπίνων δικαιωμάτων και περιβαλλοντικών ε, προτύπων. Νομίζω ότι συμφωνούμε επ' αυτού. Αυτό με οδηγεί στο εξή ερώτημα. Πώς ε, εσείς κρίνετε την εμπειρία. Δηλαδή, αν έχει υπάρξει συμβολή αυτή της συμφωνίας για την αναβάθμιση αυτών των προτύπων και στις δύο πλευρές, σε σχέση με την συμφωνία ναύτα. Γιατί αυτά τα 20 χρόνια της ναύτα εξηγούν και μεγάλες απώλειες ε, από την μεξικανική βιομηχανία και τη δυνατότητά της να ανταγωνιστεί ε, αντίστοιχη, ε, τον αντίστοιχο βιομηχανικό κλάδο στις ΕΠΑ. Επιστρέφω στα ανθρώπινα δικαιώματα. Θα σας ενδιέφερε να συμπεριληφθεί ένα τέτοιο κεφάλαιο στην αναθεωρημένη συμφωνία όπως είχε γίνει αντιστοίχως ε, με την Κολομβία και το Περού. Δεύτερο ερώτημα. Περνώ στις επενδύσεις. Στο Κοινοβούλιο έχουμε υιοθετήσει κανονισμό για την αποφυγή του ξεπλήματος του χρήματο. χρήματος. Ξέρουμε ότι χιλιάδες άνθρωποι έχουν πεθάνει, έχουν χάσει τη ζωή τους ε, στην περιοχή εξαιτίας ε, του ναρκοπολέμου. Μπορούμε μέσω οικονομικών κανονισμών να φροντίσουμε υπάρχει μάλλον περίπτωση πόροι, χρήματα που προέρχονται από εγκληματικές ενέργειες να περάσουν με κάποιον τρόπο στην ευρωπαϊκή οικονομία. Υπάρχουν νομοθετικές ρυθμίσεις για να καταπολεμήσουμε αυτό το ενδεχόμενο. Συγγνώμη, μπορείτε να συντομεύετε. Λέει ο Πρόεδρος. Και τρίτο ερώτημα. 60% του εμπορίου βάσει του προηγούμενου Γενικού Διευθυντή του ΠΟΕ Πασκαλαμή. Εφόσον είναι πολύ σημαντικός ο τομέας της ε, ε, φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής. Ε, ποια είναι η γνώμη σας για αυτό το ζήτημα σε σχέση με τις σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κύριε Μάρτιν, όχι. Εντάξει, ευχαριστώ. Από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ποιο εκπροσωπείται την Επιτροπή. Whoever is Jorgensen, yes. Thank ναι, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε τον κύριο Πρέσβη για την πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίασή του. Και εμεί από μέρου τη Γενική Διεύθυνση Εμπορίου τη ε, Κομισιόν παρακολουθούμε με ενδιαφέρον τι εξελίξει στο Μεξικό. η δουλειά που έχει γίνει στο πλαίσιο του Πάκτο México, οι μεταρρυθμίσεις ε, και η επίδραση όλων αυτών στην εμπορική πολιτική του Μεξικού είναι πράγματα που παρακολουθούμε συνέχεια. Εμείς ε, ως Κομισιόν χαιρετίζουμε και την πρόταση του Μεξικανού Προέδρου Πινιενιέτο να διερευνήσουμε τρόπους εξυγχρονισμού της ε, συμφωνίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση στο Σαντιάγκο της Χιλής ε, πέρυσι. Έχουμε προχωρήσει τη διερευνητική εργασία μαζί με το Μεξικό. Για τον πυλώνα εμπορίου έγιναν δύο συναντήσεις για το εμπόριο και τις επενδύσεις με τη σχετική υποομάδα. Εξετάσαμε όλα τα ζητήματα που προέβαλαν και τα δύο μέρη Μιλάμε για ένα τεράστιο κατάλογο θεμάτων που περιλαμβάνουν πρόσβαση στις γεωργικές αγορές, διευκόλυνση του εμπορίου, θέματα SPS, TPT, υπηρεσίες, επενδύσεις, ε, εμπόριο και επενδύσεις στην ενέργεια, ε, δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, δημόσιες συμβάσεις, ανταγωνισμός και καθώς και εμπόριο και βιώσιμη ανάπτυξη η δική μας αξιολόγηση της δουλειάς της υποομάδας είναι ότι ήταν ε, ωφέλιμη, επικοδομητική. Οι συζητήσεις ήταν παραγωγικές. Η διαδικασία έχει ληφθεί πολύ στα σοβαρά και από τα δύο μέρη. Ως αποτέλεσμα και όπως ανεφράν πολλά μέλη αποφασίσαμε να συνεχίσουμε τη διερευνητική αυτή φάση με το Μεξικό αυτή τη διαδικασία μεταξύ μας για τον εξυγχρονισμό της συμφωνίας αποφασίσαμε να ξεκινήσουμε να μελετάμε μαζί με το Μεξικό μια, ε, μια έκθεση κοινού οράματος, μια διερευνητική άσκηση, όπως κάνει πάντα η Κομισιόν όταν διερευνά τις δυνατότητες ε, ε έναρξης μιας ε, διαπραγμάτευσης για FTA με έναν εμπορικό εταίρο. Το συζητήσαμε και στην Επιτροπή Εμπορικής Πολιτικής την περασμένη εβδομάδα με τα κράτη-μέλη και λάβαμε υποστήριξη για να προχωρήσουμε σε αυτή τη διερευνητική άσκηση με το Μεξικό. Αυτή η scoping exercise, η διερευνητική άσκηση, έχει σκοπό να εντοπίσει με όσο δυνατόν μεγαλύτερη ακρίβεια τους γενικούς στόχους και τους ειδικούς στόχους καθώς και ό,τι πρέπει να επιτευχθεί συγκεκριμένα σε κάθε επιμέρους τομέα μιας πιθανής διαπραγμάτευσης. Δεν είναι λοιπόν προκαταρκτική διαπραγμάτευση. Είναι κάτι που δίνει στην κάθε πλευρά μια πολύ καθαρή εικόνα του τι επιθυμεί η άλλη πλευρά. Και αποφεύγονται έτσι δυσάρεστες εκπλήξεις κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. Υπάρχουν πολλές προκλήσεις. Πρώτη φορά διερευνάμε αναβάθμιση, εξυγχρονισμό μιας υπάρχουσας ε, συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών αλλά πιστεύουμε ότι τα αποτελέσματα θα είναι θετικά πιθανότατα. Η καλή λειτουργία της τρέχουσας συμφωνίας ε, είναι ένας ε, παράγοντας που μας οδηγεί σε τέτοιο συμπέρασμα. Η, τα πιθανά κενά και η ανάγκη εξυγχρονισμού της συμφωνίας, εάν συγκρίνουμε αυτή τη συμφωνία με τις συμφωνίες που έχουμε με χώρες όπως το Περού και η Κολομβία, καθώς και τα μεγάλα κενά σε σχέση με το ότι έχουμε συμφωνήσει με τον Καναδά και σε σχέση με ό,τι θα συμφωνήσουμε πιθανότητα με τη ΣΥΠΑ στο πλαίσιο του TTIP. Επίσης, ε, υπάρχουν ενθαρρυντικά πολιτικά σήματα από πλευράς Μεξικού και υψηλά επίπεδα φιλοδοξίας. Και αυτό είναι ένα καλό σημάδι. Για να ολοκληρώσω, κύριε Πρόεδρε, προσδοκούμε να προσβλέπουμε στη συνεργασία με το Μεξικό επί του θέματος αυτού και θα ενημερώνουμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την πρόοδο της διερευνητικής ε, άσκησης για την εξέλιξη των μελετών ε, που εξετάζουν τις επιδράσεις της σημερινής συμφωνίας αλλά και τα πιθανά ωφέλη από τον εξοχρονισμό της συμφωνίας. Επίσης θα σας ενημερώνουμε για όλες τις άλλες σχετικές πτυχές καθώς θα προχωράμε προς, μια πιθανή, προς ένα πιθανό εξυγχρονισμό της συμφωνίας. Ευχαριστώ πολύ. Πριν δώσω ξανά σε εσάς το λόγο κύριε Πρέσβη, να κάνω δύο παρατηρήσεις. Πρώτα απ' όλα κατά την άποψή μου και πρέπει να το πω δημόσια. Πρέπει οπωσδήποτε να δούμε κατά πόσο υπάρχει περιθώριο εξυγχρονισμού της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Μεξικού. Ε, έχουμε τις διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά και εσείς ανοίγετε στον ΝΑΦΤΑ, οπότε θα πρέπει να υπάρχει κάποια ευθυγράμμιση με τις ε, συμφωνίες που διαπραγματευόμαστε με τα άλλα μέρη των ΝΑΦΤΑ. Επίσης η συμφωνία μαζί σας ε, είναι λιγότερο φιλόδοξη από τη νέα γενιά συμφωνιών της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά ελπίζω πραγματικά ότι η διερευνητική άσκηση θα καταλήξει σε επιτυχή έκβαση. Επίσης, ας μην ξεχνάμε τις ε, προκλήσεις που θα δημιουργήσει αυτό για το Μεξικό, διότι αυτή η νέα γενιά συμφωνιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν τεράστιες φιλοδοξίες, περιλαμβάνουν αγαθά, υπηρεσίες, επενδύσεις, δημόσιες συμβάσεις, ε, προστασία διανοητικών δικαιωμάτων, ρυθμιστική προσέγγιση, πολλές είναι οι απαιτήσει. Και κάποια από αυτά τα στοιχεία αποτελούν ήδη και κτημένο των συμφωνιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως τα κεφάλαια για τη βιώσιμη ανάπτυξη, που περιλαμβάνουν πολύ ψηλά πρότυπα και ρήτρε ε, για περιβαλλοντικά πρότυπα. Το Μεξικό παραδοσιακά αντιτίθετο στη χρήση τέτοιων ρητρών στις συμφωνίες. Θα μπορούσε το Μεξικό να ανταποκριθεί σε αυτή την πρόκληση. Ξέρω ότι δεσμεύεστε ήδη από την ε, Βορειοαμερικανική Συμφωνία για την Ισότιμη Συνεργασία, αντίστοιχη συμφωνία με την ΑΦΤΑ, αλλά αυτό το κεφάλαιο όμως της βιώσιμης ανάπτυξης της Ένωσης μπορεί να έχει περισσότερες απαιτήσεις από τον ΑΚ. Δεύτερον, οι γεωγραφικές ενδείξεις. Οι αμερικανικές χώρες είναι αρκετά εχθρικές προς αυτή την ιδέα συνήθως. Την ευρωπαϊκή αυτή ιδέα των γεωγραφικών ενδείξεων για τα αγροτικά και διατροφικά προϊόντα θα μπορούσε να ανταποκριθεί σε αυτή την πρόκληση το Μεξικό και τρίτον να δώσω ένα παράδειγμα για τις δημόσιες συμβάσεις. Είστε ομοσπονδιακό κράτος όπως οι ΗΠΑ, ο Καναδά και ο Καναδάς και η Ευρωπαϊκή Ένωση παρεμπιπτόντως. Και φυσικά οι δημόσιες συμβάσεις έχουν διάφορες κατηγορίες, ε, ομοσπονδιακό, κρατικό, τοπικό επίπεδο. Θα μπορούσε το Μεξικό να φανταστεί να ανοίξει τις αγορές δημοσίων συμβάσεων σε ευρωπαϊκές εταιρείες. Σε αμοιβαία βάση φυσικά, ε, όχι μόνο εμείς να παρέχουμε τέτοιες υπηρεσίες. Αυτά είναι μερικά παραδείγματα συνεπειών αυτών των νέων και απαιτήσεων αυτών των νέων συμφωνιών, των εμπορικών συμφωνιών. Φυσικά το Μεξικό γνωρίζει τις προκλήσεις. Μπορείτε να μας διαβεβαιώσετε ότι είστε έτοιμοι να δεσμευτείτε. Έχετε, έχουμε πολύ λίγο χρόνο, 10 λεπτά. Κύριε Πρέσβη, ε, ε, Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω στα 10 λεπτά να τηρηθώ και να απαντήσω. Αν μου επιτρέπετε θα ήθελα να δώσω τον λόγο και στην Υπουργό Ιβόν Στίνσον που με συνοδεύει και ε, κάποιες ερωτήσεις που διατυπώσατε είναι τεχνικού χαρακτήρα, είναι διαπραγματεύτρια ουσιαστικά και θα μπορέσει εκείνη να απαντήσει. Πρώτο σχόλιο. Είναι σαφές πρέπει να το πω, έχουμε μια μικρή διαφορά όσον αφορά το τι συνέβη μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και μεταξύ ημών. Ποιος πρότεινε τον εξυγχρονισμό και την επικαιροποίηση. Αλλά αυτό δεν έχει μεγάλη σπουδαιότητα. Το σημαντικό είναι ότι βρισκόμαστε στο εγχείρημα της επικαιροποίησης με θετικό τρόπο και με καλές προθέσεις. Πρόεδρε, υπάρχουν διάφορες ερωτήσεις. Θα ξεκινήσω με τις λιγότερο γενικές, με τις γενικότερες και θα δώσω για πιο εξειδικευμένα θέματα τον λόγο στην Υπουργό να σας απαντήσει. Υπήρξαν διάφορες αναφορές στα θέματα των δικαιωμάτων του ανθρώπου και της αηφόρου ανάπτυξης. Πρώτον, πρέπει να σας πω λοιπόν ότι το Μεξικό κατά τα τελευταία 20 χρόνια πέρασε, υπήρξε σε μια διαδικασία μεταρρύθμισης βαθύτατη σε σχέση με τα θέματα εκδημοκρατισμού. Η χώρα μας εμπέδωσε γοργά και σημαντικά με αηφόρο τρόπο το κράτος δικαίου, ένα δημοκρατικό κράτος, δημοκρατικού χαρακτήρα, με μια κοινωνία δημοκρατική. Έχει λοιπόν μια δημοκρατική κοινωνία πολύ εμπεδωμένη και ολοκληρωμένη το Μεξικό σήμερα. Στα θέματα των δικαιωμάτων του ανθρώπου το ίδιο συνέβη. Δεν μπορεί να εξυγχρονιστεί και να οικοδομηθεί ένα δημοκρατικό κράτος αν δεν βασίζεται στον απόλυτο σεβασμό των δικαιωμάτων του ανθρώπου των Μεξικανών πολιτών. Και ως προς αυτό, αν παρακολουθήσετε και παρατηρήσετε όλες τις μεταρρυθμίσεις ε, τις οποίες ε, κάναμε και κάναμε λόγο για αυτές, ε, εργασιακή, εκπαιδευτική, τηλεπικοινωνιών, ένα από τα πιο σημαντικά νήματα, μύτος της Αριάδνης που διαπερνά όλα αυτά, είναι η ενίσχυση, η ενδυνάμωση των δικαιωμάτων του ανθρώπου, πολιτικών και ε, ε, δημοκρατικών, καθώς επίσης κοινωνικών, πολιτιστικών εξίσου. Το πιο σημαντικό για μας είναι να δημιουργήσουμε πολύ μεγαλύτερο ένα επίπεδο υψηλότερη ε, αναβαθμισμένης διαβίωσης, υψηλότερης ποιότητας, αναβαθμισμένης ποιότητας για τους Μεξικανούς. Θα είναι ο μόνος τρόπος για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε να αναπτυσσόμεθα και να είμαστε μια ευημερούσα αναπτυγμένη χώρα βασιζόμενη στο κράτος δικαίου, με ένα δημοκρατικό κράτος το οποίο θα διασφαλίζει απόλυτα τα δικαιώματα του ανθρώπου των Μεξικανών πολιτών. Σε σχέση με αυτό υπήρξε μια παράλληλη πολύ ενδιαφέρουσα εξέλιξη και σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά τα δικαιώματα του ανθρώπου. Μόλις τη Δευτέρα και Τρίτη είχαμε την τέταρτη σύνοδο, διμερή σύνοδο διαβουλεύσεων Μεξικού ΕΕ σε σχέση με τα θέματα των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Δέκα χρόνια είναι από τότε που ξεκινήσαμε με τη συνεργασία μας με την ΕΕ σε αυτό το θέμα. Τότε ήταν μια πολύ περιορισμένη συνεργασία στα πλαίσια της. Αυστηρά αφορούσε οικονομικά ε, θέματα όσον αφορά και την προαγωγή σχετικών θεμάτων ε, για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ο διάλογος όμως που έχουμε σήμερα, ΕΕ και Μεξικό για αυτά τα θέματα, σήμερα όχι μόνο είναι υψηλότατης ποιότητας, αλλά και πιο σημαντικό ακόμα πρόεδρε, είναι ένας διάλογος <clears throat> απόλυτα ανοιχτός, απόλυτα διαφανής και απόλυτα εγκάρσιος, οριζόντιου χαρακτήρα, διμερός, όπου αμφότερες οι πλευρές, ε, ε και Μεξικό, συμμεριζόμαστε με ειλικρινέστατο και ευθύτατο τρόπο και συζητούμε τις προκλήσεις που κάθε ένας από εμά αντιμετωπίζουμε σε αυτά τα θέματα. Και δεύτερο, εργαζόμαστε ήδη <clears throat> σε σχέση με δυνατότητες δημερού συνεργασίας και τέτοια πρότυπα που θα μας δώσουν τη δυνατότητα να επιλύσουμε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να συνεισφέρει με ουσιοδέστατο τρόπο στην ενδυνάμωση και την βελτίωση, ακόμα περαιτέρω βελτίωση το, της κατάστασης των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Αντιμετωπίζουμε σημαντικές προκλήσεις και το Μεξικό εξίσου μπορεί να συνεισφέρει σε σχέση με την ΕΕ. Να αντιμετωπίσει ΕΕ άλλες προκλήσεις εξίσου περίπλοκες υπό το ευρωπαϊκό πρίσμα, στην ίδια την ευρωπαϊκή επικράτεια. Και ένα συγκυριακά σημαντικό στοιχείο για την ποιότητα και τον πλήρη σφαιρικό χαρακτήρα για αυτά τα θέματα για τα δικαιώματα του ανθρώπου μεταξύ αμφωτέρων των πλευρών αφορά το επίπεδο, το πεδίο της προαγωγής διεθνώς των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Η παγκόσμια προώθηση προαγωγή των δικαιωμάτων του ανθρώπου σε αυτό το επίπεδο υπάρχει ένα επίπεδο κοινωνίας συμμετοχής και ε, συναλλαγής μεταξύ αμφωτέρων των πλευρών χωρίς κανένα προϊόν προηγούμενο, όπου αμφότερες οι πλευρές ενισχύουμε και προάγουμε τις δυνατότητες μας να προαχθούν σε παγκόσμιο επίπεδο τα δικαιώματα του ανθρώπου. Και αυτό αντιστοιχεί σε δύο πράγματα εντάχει. Πρώτον, είναι ένας παγκόσμιο υπεύθυνα εμπλεκόμενος στο Μεξικό και προσπαθώντας να απαντήσω στην ερώτηση της κυρίας Ευρωβουλευτού σε σχέση με την άποψη των ελίτ και τομεακά της κοινωνίας του Μεξικού σε σχέση με αυτή τη συμφωνία σύνδεσης και συσχετισμού του Μεξικού με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένωση δύσκολα η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορέσει να βρει άλλη χώρα παγκόσμια με τα χαρακτηριστικά του Μεξικού και την εμβέλεια και το εύρος και τις μεγάλες διαστάσεις του Μεξικού με τέτοιο βαθμό συγγένειας που έχει το Μεξικό με εσά σε όλα αυτά τα θέματα, πολιτιστικά και πολιτισμικά, αξιών και αρχών, οράματος. Είμαστε δημοκρατικά κράτη, είμαστε κράτη και έθνη που πιστεύουμε στα δικαιώματα του ανθρώπου και την ελευθερία και προάγουμε την ελευθερία ελευθερία με κάθε τρόπο. Αυτό είναι εκείνο που μας οδήγησε ώστε για μας το Μεξικό πιο φυσικός εταίρος του υπό οποιαδήποτε πρίσματα ε, και σε σχέση πέρα από το γεωγραφικό θέμα να είναι ο πιο ε, συγγενής εταίρος η Ευρωπαϊκή Ένωση. Το, η απάντηση λοιπόν είναι ένα καταφατικό ναι, απόλυτο ναι. Η κοινωνία του Μεξικού, το Μεξικό, οι πολίτες, η κυβέρνηση θέλουμε να προχωρήσουμε σε σχέση με αυτές τις διαπραγματεύσεις. Για την ΑΦΤΑ και την ε, Διατλαντική Συμφωνία Εμπορίου και Επενδύσεων ο συσχετισμός με την TTIP πρέπει να ερμηνευτεί με το συμφέρον ή όχι σε σχέση σχέση με τον Καναδά και τον Μεξικό υπό το εξή πρίσμα. Η ναύτα ένα από τα πιο σημαντικά αποτελέσματα που είχε είναι ένας βαθμός ολοκλήρωσης στη Βόρεια Αμερική σε υψηλότατο βαθμό. Υπάρχουν οικονομικοί τομείς, βιομηχανικοί τομείς στη Βόρεια Αμερική που <clears throat> έχουν ολοκληρωθεί και έχουν ενταχθεί αυτό που διαπραγματεύεται, ε, ε, διαπραγματεύονται η ΙΠΑ, ο Καναδάς, το Μεξικό και μεταξύ ημών και της ΕΕ, όλα αυτά έχουν επιπτώσεις στον υπόλοιπο κόσμο. Υπό αυτό το πρίσμα πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε. Δεν θέλω να πω ότι θέλει το Μεξικό να γίνει τμήμα αυτής της διαπραγμάτευσης, αλλά έχουμε κάθε ενδιαφέρον να προχωρήσουν αυτές οι διαπραγματεύσεις και τις παρακολουθούμε εκ του σύνεγγης, διότι αποτελούμε μέρος ενός, ε, μιας πολύ ολοκληρωμένης ενωμένης αγοράς με τις ΗΠΑ. Για την ερώτηση αν δίνει θετικά μαθήματα η ναύτα υπό το φως και των διαφορών, της μεγάλης διαφοράς ε, σε σχέση με την ανάπτυξη μεταξύ των δύο χωρών πριν από 20 χρόνια, η απάντηση είναι πολύ θετική. Είναι ένα θετικό ναι. Πρώτα απ' όλα η ναύτα δεν ήταν μόνο απλά ένα, ε, μια συμφωνία που απελευθέρωσε τις εμπορικές σχέσεις στη Βόρεια Αμερική. Είναι μια συμφωνία που όθησε το Μεξικό να εξυγχρονιστεί και να επικαιροποιηθεί. Μας υποχρέωσε να εξυγχρονίσουμε τα θεσμικά μας όργανα, να εξυγχρονίσουμε την νομοθεσία μας. Μας υποχρέωσε να αναβαθμίσουμε τις προδιαγραφές και τις διατάξεις με τις οποίες λειτουργούσαμε με πολύ σημαντικό τρόπο. Χωρίς την παραμικρή αμφιβολία υπέστησαν πλήγματα πολλές επιχειρήσεις από αυτό το άνοιγμα, διότι δεν είχαν συνηθίσει και προσαρμοστεί να ανταγωνίζονται σε μια ανοιχτή αγορά και με αυτές τις πιέσεις. Μέσα σε όλα αυτά τα χρόνια το αποτέλεσμα είναι πολύ ξεχωριστά θετικό. Μέσα σε 20 χρόνια από διαμαρτυρίες και διακόπτουν στην αίθουσα χωρίς μικρόφωνο. Χωρίς μικρόφωνο. Σας ευχαριστώ λέει ο πρέσβης. Το εμπόριο του Μεξικού εδώ και 20 χρόνια πριν υπογραφή είναι αυτά ήταν, 500, ε, ήταν 50 δις δολάρια και 20 χρόνια μετά σε θετικό βαθμό χάρη στην ναύτα είναι 800 δισεκατομμύρια δολάρια αυτό το εμπορικό, ο εμπορικός όγκος και είναι μεταποιημένα προϊόντα πάπου παράγονται στο Μεξικό. Ναι, λίγο χρόνο σας και έχετε εξαντλήσει το χρόνο, πρέσβη. Εντάξει, ολοκληρώνω και δίνω τον λόγο την Υπουργό, ώστε σε τεχνική ερώτηση να μπορέσει να αποσαφηνίσει κάποια πράγματα. Παρακαλώ, έχετε τον λόγο εσείς κυρία. Μάλιστα σας ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία να είμαστε εδώ ανάμεσά σας και να μπορέσουμε να πούμε δύο λόγια για τη χώρα μας. Πράγματι βρισκόμαστε σε αυτή τη διαδικασία της ε, εξέτασης ε, και προώθησης των επιπέδων ε, ανάπτυξης των σχέσεών μας μεταξύ ΕΕ και Μεξικού είχαμε ήδη δύο συνεδριάσεις και τώρα ακριβώς εργαζόμαστε για την προώθηση αυτού του ολοκληρωμένου οράματος. Όπως κάθε διαρευνητική διεργασία όλα τα θέματα που είναι στο τραπέζι όλα θα εξεταστούν και θα συζητηθούν. Και όταν θα έχει ξεκινήσει η διαδικασία διαπραγματεύσεων τότε θα αποφασίσουμε ποια από αυτά τα θέματα και με ποιες ρήτρε μπορούν να συμπεριληφθούν και με ποιο τρόπο. Σε αυτή τη συγκεκριμένη στιγμή μπορούμε να απαντήσουμε μόνο για το θέμα όσον αφορά το κεφάλαιο της αηφόρου ανάπτυξης. Προφανώς θα υπάρξει ένα τέτοιο κεφάλαιο. Ποιες θα είναι οι ρήτρες του, αυτό θα το δούμε στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης και θα το διαμορφώσουμε σε σχέση με τις προτάσεις όσον αφορά την ΕΕ και το Μεξικό. Για την, το μηχανισμό επίλυσης διαφορών, το μηχανισμό τον έχει συμπεριλάβει σε σχεδόν όλες τις συμφωνίες και συνθήκες του και έχουμε συμφωνίες με 16 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε ήδη αυτό το μηχανισμό λοιπόν από πλευράς μας. Νομίζω ότι στη στιγμή της διαπραγμάτευσης εμείς θα συζητήσουμε όταν έρθει η ώρα με την ΕΕ τις δυνατότητες να υπάρξει ένας μηχανισμός προστασίας προφανώς των επενδύσεων και αν είναι σκόπιμο ή όχι επίσης να υπάρξει αυτή η διαιτησία, επιδιαιτησία μεταξύ διαιτητικών ε, ε, σωμάτων ή φορέων που θα μπορούν να συζητήσουν και να διασαφηνίσουν συγκεκριμένα θέματα μιας παραβίασης ή παράβασης. Το θέμα για τη Συμφωνία για το Ελεύθερο Εμπόριο θέλω να το προσθέσω η ναύτα ήταν πολύ σημαντική για μας. Πριν από 20 χρόνια δεν μπορούσε κανείς να φανταστεί ότι μια οικονομία όπως η μεξικανική οικονομία θα μπορούσε να έχει μια συμφωνία ελεύθερου εμπορίου με μια οικονομία της κλίμακας όπως ε, της κλίμακας των ΗΠΑ και του Καναδά. Αυτή τη στιγμή εδώ και 20 χρόνια η χώρα μου άλλαξε άρδιν όπως το εξέφρασε και ο πρέσβης και υπό, υπό, όρου οικονομικούς όρους έχουμε σημειώσει πολύ μεγάλη πρόοδο και με τις μεταρρυθμίσεις, τις ε, επικαιροποιημένες ε, επι, ε, μεταρρυθμίσεις αυξάνουμε την ανταγωνιστικότητα και την παραγωγικότητα. Ανταγωνιστικότητα να έχουν την ευκαιρία να έχουν θέση απασχόλησης οι Μεξικανοί και για τα ζητήματα βίας, ληστιών, κλοπών, όλα αυτά τα προβλήματα θα μπορούν να επιληθούν όταν οι νέοι Μεξικανοί θα έχουν μια θέση απασχόλησης, θα έχουν κάποια έσοδα που θα είναι βελτιωμένα σε σχέση με τη σημερινή του κατάσταση. Για το θέμα του Ευρωβουλευτή Βιτάλ Μορέιρα, είμαστε έτοιμοι να διαπραγματευτούμε εμεί. Έχουμε 10 συνθήκες συμφωνίες με 45 χώρες. Εμείς με μετά από την ΑΦΤΑ, μετά από τη Συμφωνία Ελευθέρου Εμπορίου για τη Βόρεια Αμερική, έχουμε αναπτύξει σχέσει με όλε τι χώρε του κόσμου. Είμαστε πρόθυμοι λοιπόν να διαπραγματευτούμε, να καθίσουμε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και να δούμε τα επίπεδα φιλοδοξιών που υπάρχουν και να δούμε ποια θα είναι η συναλλαγή. Μια και μια Συμφωνία Ελευθέρου Εμπορίου, όπω έχει αναφερθεί, είναι ένα θέμα win-win κερδίζουν και οι δύο. Δεν είναι μηδενικού αθροίσματος παιχνίδι. Ευχαριστώ. Πράγματι λέει ο κύριος Μωρέ. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Πρέσβη, ευχαριστούμε πολύ κύριε Ακούριε για την παρουσία σας εδώ. Μπορούμε τώρα να προχωρήσουμε στο επόμενο θέμα τις ψηφοφορίας. Σας δίνω ένα λεπτό για να προετοιμάσετε τις ε, λίστες ψηφοφορίας, τις κάρτες σας. Δεν είναι και πολλά, μόνο τρία είναι τα θέματα. Πρώτον, έγκριση της συμφωνίας μεταξύ των δύο συνομοθετών για ε, το σύστημα αδειών για τις εισαγωγές ξυλίας στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Γιούλιου Βίνκλερ. Πρόκειται για την τελική ψηφοφορία. Άρχεται. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται ομοφόνος. Συγχαρητήρια. Μετά. Για τα είδη διπλής χρήσης και πάλι πρόκειται για έγκριση της ε, συμφωνίας μεταξύ Συμβουλίου και Κοινοβουλίου, τελική ψηφοφορία, έναρξη ψηφοφορίας. Πέρας. 22 ψήφοι υπέρ, 0 κατά, 3 αποχές, εγκρίνεται λοιπόν με συντριπτική πλειοψηφία. Συγχαρητήρια στον κύριο Φιέλνερ. Σημείο 16. Τελωνιακή δασμή για την Ουκρανία. Συγητής ο κύριος Ζαλεύσκη. Ο κύριος Ζαλεύσκη, ευχαριστώ πρόεδρε. Γιατί ήθελα να πάρω το λόγο επειδή Υπάρχει τροπολογία που αναφέρεται στα ανθρώπινα δικαιώματα. Να σας ενημερώσω ότι αύριο η κυβέρνηση της Ουκρανίας ε, θα υπογράψει το πολιτικό τμήμα της ε, συμφωνία Σύνδεση, όπου δεσμεύεται να διασφαλίσει την τήρηση των ανθρωπινών δικαιωμάτων. Και νομίζω ότι έτσι ε, καλύπτονται όλες οι προσδοκίες μας. Επομένως, Σας ε, καλώ λοιπόν να μην στηρίξετε την τροπολογία αυτή. Εντάξει, σαφή όλα αυτά. Ας ψηφίσουμε την τροπολογία 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ας ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Τροπολογία 2. Άρχεται πέρας απορρίπτεται. Τροπολογία 2, να υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Προ... Ψηφίζουμε την πρόταση της Επιτροπής ως έχει, άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται με 22 ψήφους υπέρ. Δύο κατά και μία αποχή. Ε, σχέδιο ψηφίσματος, άρχιτε ψηφοφορία, πέρας. Το ίδιο αποτέλεσμα, 22 υπέρ, 2 κατά, μία αποχή. Συγχαρητήρια στον εισηγητή. Φτάνουμε στο τέλος ε, των ψηφοφοριών. Uh, this uh, voted in plenary. Λοιπόν, θα ψηφιστεί την Ολομέλεια στην πρώτη σύνοδο του Απριλίου. Σημείο 17. Όσοι θέλουν να αποχωρήσουν, ας το πράξουν. Οι υπόλοιπες καθίσουν. Πρόεδρε, επί της διαδικασίας. Ναι, πραγματικά επί της διαδικασίας. Δεν θέλω να φανώ μικροπρεπής, όμως έχουμε λάβει τις κριτικές από άλλα κόμματα ε, σε ό,τι φορά την ε, Επιτροπή και εδώ βλέπουμε ότι ε, άλλο μέλος, αναπληρωματικό μέλος άλλης πολιτικής ομάδας έχει κρύψει το καρτελάκι μου και έχει καθίσει σε ε, στη θέση κανονικού μέλους ε, αντί να καθίσει στη θέση της και δεν ξέρω αν αυτό είναι σωστό ή όχι. Ο Πρόεδρος, ναι, πρόκειται για συνωμοσία κατά της πολιτικής σας ομάδας. Ναι, παρακαλώ μην το κάνετε. Okay, <laughs> Item 7. Σημείο 17. Η κατάσταση όσον αφορά τις συμφωνίες οικονομικής εταιρικής σχέσης. Συνήθως ε, αποκαλούνται ΕΠΑΣ. Όπως ξέρετε, έχουμε υιοθετήσει κανονισμό ε, πρόσβαση στην αγορά που θεσπίζει προθεσμία για την σύναψη των διαπραγματεύσεων ε, και ολοκλήρωση διαπραγματεύσεων με αυτές τις ομάδες για την αντικατάσταση ε, των υφιστάμενων εμπορικών προτιμήσεων με εμπορικές συμφωνίες. Η προθεσμία αυτή είναι η 1η Οκτωβρίου 2014. Βεβαίως, καθώς ε, ολοκληρώνεται σιγά σιγά η κοινοβουλευτική μας πρέπει να να γνωρίζουμε πώς έχει η κοινοβουλευτικη μα θητεια πρεπει να γνωριζουμε πω εχει η κατασταση Αλεξάνδρα Γαλίνα έχει τον λόγο γιατί ε, είναι και αυτή που τα γνωρίζει καλύτερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πολύ καλή αυτή εισαγωγή. Ναι, πώς έχει η κατάσταση. Να σας δώσω μια επισκόπηση. Ουσιαστικά πρέπει να μιλήσουμε για την εφαρμογή και τις διαπραγματεύσεις, γιατί τα δύο αυτά συνδέονται στενά. Σε ό,τι αφορά το επίγον τμήμα των διαπραγματεύσεων, θα γίνει συνεδρίαση με τους ε, εταίρους EAC την επόμενη εβδομάδα, όπως ξέρετε, με την ε, κοινότητα Ανατολικής Αφρικής, ε, για να ολοκληρώσουμε την εξέταση των λίγων αυτών ζητημάτων που μας απομένουν. Από 7 μένουν και από αυτά τα 3 είναι τα πιο σημαντικά κάποιες ρήτρες, ε, η ρήτρα μη εκτέλεσης που συνδέεται με το άρθρο 96 και το καθεξής. Τα υπόλοιπα τέσσερα σημεία ε, είναι ίσονο σημασία. Για το ΣΑΝΤΕΚ, για την κοινότητα και την ανάπτυξη της Μεσευρινής Αφρικής, θα γίνει ε, ακόμα μία προσπάθεια ολοκλήρωσης αυτής της EPA, Συμφωνίας Οικονομικής Εταιρικής Σχέσης, και μετά Πρέπει να πω ότι το πιο σημαντικό εδώ είναι η εξαγωγική φόρη ή ίσως συνδέονται και με άλλα ζητήματα όπως ε, οι διασφαλίσεις. Από όσο γνωρίζουμε εμείς, ε, άλλα ζητήματα όπως η πρόσβαση στην αγορά και η γεωργία, η πρόσβασή μας δηλαδή στην Νότια Αφρική και η πρόσβαση της Νότιας Αφρικής στην Ευρώπη, συγγνώμη που το λέω τόσο κατονομάζω τη χώρα, αλλά είναι σαφές για όλους μας, νομίζω ότι όλα αυτά κινούνται ε, ομαλά. Ας συνεχίσουμε λοιπόν ε, αυτή τη διαδικασία. Λοιπόν, αυτές είναι οι δύο περιοχές όπου υπάρχουν πραγματικές διαπραγματεύσεις ε, που ίσως ε, να ολοκληρωθούν μέχρι την προθεσμία που έχουμε θέσει. Για τις υπόλοιπες διαπραγματεύσεις δεν θέλω να σας κουράσω. Ε, κινούνται πιο αργά, υπάρχει μάλλον μια κοιλιά, αν το θέσω έτσι, γιατί για την ε, Κεντρική Αφρική δεν υπάρχει άμεσος αντίκτυπος γιατί εκεί το ενδιαφέρον είναι η εφαρμογή. Σκεφτόμουν προηγουμένω που βρισκόμασταν το 2009, όταν ξεκίνησε αυτή η κοινοβουλευτική θητεία και πρέπει να πω ότι ε, ήμουν ιδιαίτερα ευγνώμων προς εσάς, προς όλους εσάς, γιατί νομίζω ότι έχει αλλάξει πολύ σημαντικά το τοπίο. Αν θυμάστε τότε δεν ε, είχαμε και πολλά σε ό,τι αφορά την εφαρμογή. Υπό αυτή την κοινοβουλευτική θητεία είχαμε και περάσαμε τρεις ε, ιδιαίτερα αμφιλεγόμενες ε, ε, EPAs. Μιλώ για την ενδιάμεση συμφωνία για τον Ειρηνικό, για την Κεντρική Αφρική και για την Ανατολική και Νότια Αφρική. Σας ευχαριστώ λοιπόν όλους γιατί αυτό σημαίνει ότι η εφαρμογή μπορεί να ξεκινήσει με ε, συνένεση. Σε κάποιες ε, περιοχές αυτό έχει ήδη ξεκινήσει στις δύο πρώτες περιπτώσεις. Νομίζω ότι το τοπίο έχει αλλάξει δραματικά γιατί όπως είπατε και εσείς έχουμε εισαγάγει αυτό το στοιχείο που αλλάζει τους όρους του παιχνιδιού. Ήταν δύσκολο για όλους μας, όμως οι προθέσεις ε, ήταν θετικές. Θέλουμε επιχειρηματική δραστηριότητα, θέλουμε συνεχιζόμενη συνεργασία με τους εταίρους μας. Γι' αυτό και το θέτουμε σε μια εύρωστη βάση, για να μην είναι εύκολο θύμα επίθεσης από άλλους. Εφαρμογή λοιπόν, συνεχίζουμε την ίδια προσπάθεια. Ήδη είχαμε τρεις συνεδριάσεις της Επιτροπής ε, που χειρίζεται αυτά τα ζητήματα, συν δύο συνεδριάσεις του Συμβουλίου. Συνεχίζουμε τώρα με την ε, ε, αναθεώρηση. Κινούμαστε ταχύτατα και ελπίζω να μπορέσω να σας ενημερώσω και πάλι. Σε ό,τι αφορά τον ειρηνικό, ξέρετε ότι το PNG είναι μια μεγάλη επιτυχία. Δεν χρειάζεται να πω και πάλι ότι πρόκειται για κέρια σημασίας ε, μέτρο και συμφωνία και αυτό θα ισχύσει και για οποιαδήποτε άλλη χώρα της περιοχής θα το κυρώσει. Θα σταματήσω εδώ για να ακούσω και τα ερωτήματά σας, αλλά και πάλι να σας ευχαριστήσω για όσα κάνατε, ακόμα και με πολύ δύσκολες αποφάσεις όπως ήταν κάποιες φορές, όπως η τροποποίηση του κανονισμού πρόσβαση στην αγορά, που ουσιαστικά δεν θέτει τέλος στις διαπραγματεύσεις. Διευκρινίζω ότι οι διαπραγματεύσεις πάντα συνεχίζονται, δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Το θέμα είναι πώς φτάνουμε όσο εκεί με την συνέχιση των προτιμήσεων μετά την προθεσμία. Και εκεί οι εταίροι μας έχουν το δικό τους, ε, τη δική τους προσέγγιση. Σας ευχαριστώ πολύ. Ε, Ευχαριστούμε πολύ. Ας ακούσουμε τώρα τους δικούς μας συγγετές αυτής της Επιτροπής των διαφόρων ομάδων ΑΚΕ. Ας ξεκινήσουμε την κυρία Κασπάρη που ασχολείται με την ομάδα των χωρών της Ανατολικής και της Μεσημβρίνης Αφρικής. Αξιότιμε Πρόεδρε, νομίζω τα όσα αναφερθήκαν είναι αυτά τα οποία ελπίζουμε σε σχέση με εκείνη την ημέρα των εκλογών που φτάνει όλο και πιο κοντά. Θα ήμουν ευγνώμων αν το 2014 καταλήγαμε σε ένα αποτέλεσμα και θα ήμουν ευγνώμων αν η Επιτροπή και για τα, τους όσους ε, εμπλέκονται που Είμαι βέβαιος ότι θα το προσπαθήσουν. Αν τώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον χρόνο πριν από τις εκλογές ε, μέχρι το καλοκαίρι, μέχρι τον Οκτώβριο, Νοέμβριο, να μην ε, ε, σταυρώσει τα χέρια, να καταλήξουμε σε ένα αποτελέσματα. Έδειξε το Ευρωκοινοβούλιο τις καλές του προθέσεις και συνεισφέραμε ώστε η μεταβατική περίοδος να επεκταθεί. Ξέρουμε τα προβλήματα που υπήρχαν και είναι σημαντικό οι χώρες που καλούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καταλήξουν σε ένα αποτέλεσμα. Δεν θα υπησέθω σε λεπτομέρειες. Κρίμα είναι το ότι δεν τα καταφέραμε. Το θέμα αυτό το μας έχει απασχολήσει στην ε, Κοινοβουλευτική μας Επιτροπή. Θα έπρεπε αυτό το χρονικό διάστημα μετά τις εκλογές να το εγγράψουμε στην ημερήσια διάταξη ώστε να προχωρήσουμε και κάτι να γίνει. Ευχαριστώ. Um... Christopher Fiala is not there. He is responsible for Western Africa, West Africa, where a breakthrough was achieved with ECOWAS. Um, what, what are the Ποια είναι τα εκκρεμή ζητήματα όσον αφορά τη συμφωνία Έχω ακούσει κάποιες αμφιβολίες ότι φουσκώνουμε υπερβολικά τις φιλοδοξίες μας ε, για τα επόμενα 20 έτη. Ότι είναι κάπως υπερβολικές Dave Martin για την Κεντρική Αφρική, τον Ειρηνικό. Θα πρέπει να σας τα δώσουμε όλα σε εσά αφού έχετε τόσο μεγάλη επιτυχία. Θα μπορούσα να το δεχτώ, λέει ο κύριος Μαρτίν. Έχω πολύ λίγες ερωτήσει. Όσον αφορά την αναθεώρηση Κάριφων, είναι ενδιαφέρον το χρονοδιάγραμμα. Τον Οκτώβριο δηλαδή όταν θα επανέλθουμε θα μπορέσουμε να δούμε την αναθεώρηση και πρέπει να δούμε επίσης ε, την έκταση που προγραμματίζει η Κομισιόν ε, κοιτάμε να δούμε σε ποιο βαθμό έχει υλοποιηθεί ή κατά πόσο βοηθά τις ε, οικονομίες της Καραϊβικής και κατά πόσο υπάρχουν θετικά και αρνητικά ε, παραδείγματα από την ελευθέρωση των ε, σχέσεων με τις χώρες της Καραϊβικής. Ναι, αυτή είναι μια ιστορία επιτυχίας των ΣΟΕΣ. Όποιος την να μιλήσει με ανθρώπους από την Παπουανέου ή η Κομισιόν θα γνωρίζει ότι στο Κοινοβούλιο αυτό η Επιτροπή Αλίας ιδιαίτερα αλλά και το Ισπανικό Λόμπι αν μπορώ να το πω έτσι αντιτίθετο σε αυτή την συμφωνία γιατί έλεγαν ότι θα πλήξει τα συμφέροντα των Ισπανικών ε, ε, βιομηχανιών αλλά το αποτέλεσμα ήταν το αντίθετο βοήθησε τις ε, εταιρείες κονσερβοποίησης τόνου στην Ισπανία Καλό είναι αυτό να γνωρίζουμε ότι βοηθούνται αφότερε πλευρέ συμφωνία. Τώρα, όσον αφορά την Κεντρική και τη Μεσαιβρινή Αφρική, δεν ξέρω αν έχω να κάνω κάποιο σχόλιο για την Κεντρική Αφρική. Ευχαριστούμε. Ο κύριο Στέρντι. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστούμε την Επιτροπή. Χαίρομαι ιδιαίτερα που ακούω τα όσα είπατε ότι η κατάσταση βελτιώνεται. Ευχαριστώ που ήσασταν πάντα ειλικρινεί μαζί μα. πολύ ωφέλιμο η Κομισιόν να είναι τόσο ειλικρινής μαζί μας ε, επί αυτών των ζητημάτων. Θα ήθελα να διευκρινίσουμε το εξής. Είπατε ότι η Γεωργία έχει επιληθεί. Υπήρξε το μαύρο πρόβατο των περισσότερων διαπραγματεύσεων και χαίρομαι ιδιαίτερα και γνωρίζω μια, ιδιαίτερη χώρα, μια συγκεκριμένη χώρα που δημιουργούσε ιδιαίτερο πρόβλημα την οποία αναφέρατε. Επίσης αναφέρατε ότι υπήρχε ένα πρόβλημα με τους, ε, με τους δασμούς ε, επί των εξαγωγών. Μπορείτε να πείτε γιατί δασμούς πρόκειται, είναι δασμοί επιγεωργικών προϊόντων, όχι, βιομηχανικών προϊόντων που ε, προκύπτουν από την ομάδα SADC. Το κατά πώς το καταφέρουμε να τα αυτά σε αυτό το κοινοβούλιο, αυτή είναι η άλλη ερώτηση, επειδή εγώ ήμουν εισηγητής για τις ΣΟΕΣ ε, αρχικά πριν από πολλά χρόνια. Ήθελα να δω να ολοκληρώνεται το θέμα πριν το τέλος της θητείας αυτού του κοινοβουλίου, αλλά ευχαριστούμε Ρόμπερτ. Τέλος Χέλμοντ Σόλτς για την κοινότητα Ανατολικής Αφρικής. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ θα είμαι λιγάκι πιο επικριτικός για όλες τις ΣΟΕΣ, αλλά και για τη δική μου περιφέρεια. Πιστεύω ότι μέχρι στιγμή η εικόνα έχει ως εξή. Υποδιαιρούμε τις περιφέρειες όπου συνάπτουμε ΣΟΕΣ. Δηλαδή έχουμε την Κάριφόρμ και όλες τις υπόλοιπες. Μπορείτε να δώσετε ένα συγκεκριμένο παράδειγμα κομισιών όπου όλες οι εταίρες χώρες μαζί συνάπτουν την ΣΟΕΣ και αν όχι γιατί όχι. Τέλος, όσον αφορά την κοινότητα Ανατολικής Αφρικής, παραμένει το ερώτημα του τι θα γίνει με την Κένια και την Αμίμπια μετά από την 1η Οκτωβρίου. Κατά πόσο θα μπορέσουμε δηλαδή να συνεχίσουμε με αυτό ή με το επόμενο κοινοβούλιο. Πώς θα αντιμετωπίσουμε το ζήτημα και τι πιθανότητες έχει η Ναμίμπια να διατηρήσει το θέμα των δασμών στις εξαγωγές ως ευκαιρία να αναπτυχθεί ως οικονομία και τι γίνεται με την Κένια κατά πόσο διαφέρει η κατάσταση εκεί και αν έχουν τη δυνατότητα να ε, συνάψουν αυτή τη ΣΟΕΣ. Δέιβιντ, ε, ζητήστε το λόγο. Συμφωνώ με τον Χέλμοντ. Ε, ήθελα να τονίσω τώρα για την Cariform. Το έχουμε συζητήσει πολλές φορές Κατά τη δική μου αξιολόγηση, κομμάτι της μεγάλης επιτυχίας ε, για την Καριφόρμου ήταν ότι όλες οι χώρες ε, συνεργαστηκαν στενά, περισσότερο από ό,τι στην ιστορία τους ποτέ. Και η ΣΟΕΣ αποτέλεσε κινητήριο δύναμη γι' αυτό. Η γραμματεία Καριφόρμ αποτελεί ένα εξαιρετικό παράδειγμα γραμματείας που υποσ... Ε, υπόδειγμα για τη ΣΟΕΣ γενικότερα. Η συνεργασία δεν είναι ποτέ τέλεια, αλλά είναι πολύ ψηλότερο επίπεδο από ό,τι ήταν ποτέ σε μια τόσο ξεχωριστή περιφέρεια όπως ε, η Καραϊβική ε, λειτουργήσε πάρα πολύ καλά στην ολοκλήρωση μεταξύ αυτών των χωρών. Άλλα μέλη της ε, Επιτροπής, πέρα των εισηγητών. Ναι, παρακαλώ κύριε Σόλτς, όχι. Για να διευκρινίσω είπα εκτός της Καριφόρμ. Αναγνωρίζω δηλαδή ότι η Καριφόρμ ε, επέτυχε αυτά που έπρεπε, αλλά όχι άλλες. Ε, επιτρέψτε μου λοιπόν ως πρόεδρος της Επιτροπής, καθώς ήταν στο τέλος της να συμφωνήσω με την Κομισιόν. Ήταν πολύ θετικές εξελίξεις σε σύγκριση με την κατάσταση το 2009. Εγώ υποστηρίζω τις ΣΟΕΣ ε, για τρεις λόγους. Πρώτον, βοηθούν να ευθυγραμμίζεται η κατάσταση με τον ΠΟΕ και να τερματίζεται μια παράνομη κατάσταση όπου εμείς εξακολουθούμε να δούμε προτιμησιακά καθεστώτα πέραν της γραμμής που έχουν χαράξει αυτοί στο πλαίσιο του ΠΟΕ. Δεύτερον, για την υποστήριξη της περιφερειακής ολοκλήρωσης των χωρών ΑΚΕ διότι περισσότερες από αυτές τις συμφωνίες, όλες τους ε, αποσκοπούσαν να είναι ε, διαπεριφερειακές συμφωνίες και όχι με επιμέρους ε, χώρες. Και τρίτον, γιατί αυτή είναι μια νέα προσέγγιση όσον αφορά τις οικονομικές μας σχέσεις με τις χώρες ΑΚΕ. Αντί για αναπτυξιακή βοήθεια, έχουμε ενεργό συμμετοχή στην ανάπτυξη μέσω του εμπορίου. Για αυτούς τους λόγους, κατά την απόψη μου, αιτιολογείται αυτή η άσκηση. Και θα ήθελα να συγχαρώ την Επιτροπή και να ε, εκφράσω την υποστήριξή μας. Ε, σαν τρέχετε τον λόγο. Ευχαριστούμε εμείς ε, ιδιαίτερος από τη δική μας πλευρά. Κάποιες ερωτήσεις ήταν πολύ ενδιαφέρουσες. Ε, μπορώ να σας δώσω κάποιες παρα, παραπληροφορίες για την Ε, Ήθελα να απαντήσω αμέσως. Πρέπει να δείτε τη συνολική συμφωνία. Κάποιοι με ρωτούν ε, τι είναι αυτά τα νούμερα που βλέπουμε. Αν δείτε τη συμφωνία σε βάθος θα δείτε ότι υπάρχει μια πολύ καλή ρήτρα για τους δασμούς, ε, για τις εξαγωγές. Βασίζεται στην ιδέα ότι δεν είναι μέσω τέτοιοι δασμοί πρόωθησης ανάπτυξης και πλούτου σε μια χώρα. Μπορώ να δώσω και άλλα τέτοια παραδείγματα και αν το επιθυμείτε μια μέρα μπορούμε να οργανώσουμε και μια τεχνική ακρόαση επί του θέματος. Θα ήθελα να αναφερθώ στους δασμούς επί των εξαγωγών και την ερώτηση για την ομάδα Σάντακ. Γιατί είναι σημαντικό να καταλάβετε τι συμβαίνει. Όπως γνωρίζετε η Νότια Αφρική δεσμεύτηκε ώστε να μην έχει δασμούς στις εξαγωγές, ε, ουσιαστικά παγώσαμε την κατάσταση. Όταν συνάψαμε την TDCA, αυτό που συνέβη ήταν πολύ ενδιαφέρον. Εμείς ήμασταν έτοιμοι να ακολουθήσουμε μια πολύ ευέλικτη προσέγγιση για όλες τις χώρες, συμπεριλαμβανομένες της Ναμίμπια, χορηγώντας σε όλους τη δυνατότητα να επιβάλλουν δασμούς για έσοδα, για τη βιομηχανική ανάπτυξη. Ο κατάλογος ε, είναι τεράστιος και δεν ε, περιορίζει τη δυνατότητα οποιασδήποτε χώρας να επιβάλλει φορολογία. Για την Νότια Αφρική θέλαμε να αποφύγουμε να επιβάλλουν τέτοιους φόρους για την βιομηχανική ανάπτυξη. Αυτή είναι η διαφορά μεταξύ μας και ε, μας εμποδίζει να καταλήξουμε συμφωνία. Το αστείο είναι και όπως αναφέρεται την Ναμίμπια, η Ναμίμπια έχει τον πιο ευελίκτο κανονισμό ουσιαστικά υπερασπίζεται την Νότια Αφρική. Μάχεται αντί αυτής. Γιατί το λέω αυτό διότι όταν αναφέρει κανείς την Κένια ή την Ναμίμπια ως ε, ανησυχητικές περιπτώσεις, εγώ πρέπει να πω ότι δεν συμφωνώ. Η Ναμίμπια είναι μια χώρα μεσαίων προς υψηλών ε, εισοδημάτων που δεν ε, υπόκειται σε καθεστώς ε, προτιμησιακό Ξέρετε, οι χώρες αυτές δεν θα υπογράψουν τις 27 συμβάσεις. Χορηγούμε ε, αφορολόγητο χωρίς ποσοστό σε αυτές τις φορές ε, και θα δούμε κατά πόσο μπορεί να χρησιμοποιηθεί το εμπόριο για να υπερασπίσουμε τις αξίες μας σε όλη την γάμα. Αφήντα το πλάι λοιπόν πολιτικές αποφάσεις που δεν με αφορούν, Πιστεύω σίγουρα ότι αυτή τη στιγμή η Κένια βρίσκεται σε μία, μπροστά σε μια διπλή επιλογή. Έχουν ένα εμπορικό σύστημα όπου η Ινδία ε, είναι ο μεγαλύτερος εταίρος. Το 3% των εξαγωγών τους, και αυτό είναι μικρό κλάσμα, επηρεάζεται από αυτό. Και δεν είναι τεράστιο ποσοστό αυτό, γιατί λέω 3% γιατί υπάρχει το γενικό πρωτοσημιακό καθεστώ, υπάρχει η γένεια, ε, είναι μια κανονική χώρα που εντάσσεται στο GSP και καλύπτει ότι οι περισσότερε εξαγωγέ τη. στο κλάσμα που δεν θα καλύπτεται μετά από την 1η Οκτωβρίου θα είναι αυτό το 3% με δασμού που δεν είναι υπερβολικοί. Πρέπει σταθμισμένα δηλαδή να προσεγγίζουμε την κάθε περίπτωση. Θεωρώ ότι μια χώρα όπως η ακτή ελεφαντοστού έχει πολύ περισσότερα να χάσει αν δεν έχει ΣΟΕΣ από την Κένια. Η Κένια το ξαναμελετά. Πολιτικά λοιπόν πρέπει να, επιλε... να σεβαστούμε τις επιλογές τους. Εάν θέλουν να συμμετάσχουν, όπως σας είπα, ε, οι φραγμή μεταξύ μας ε, είναι ζητήματα στα οποία δεν έχουμε μεγάλο περιθώριο λιγμού. Δεν μπορώ να έρθω σε αυτό το κοινοβούλιο με μία σώση που να μην έχει ρήτρα μη εκτέλεσης. Δεδομένων των προσφάτων ετοιμάτων για την ομοφοβία και τα λοιπά στοιχεία, θέλω να πω, εμείς έχουμε τις δικές μας αξίες, έχουμε μια εμπορική πολιτική αλλά και αξίες. Κατά την απόψή μου λοιπόν, πρέπει να ανησυχούμε για την προθεσμία για ορισμένε χώρες. Έχουν κάνει αυτές τις χώρες ό,τι χρειαζόταν. Στην ΕΚΟΒΑΣ έχουμε ολοκληρώσει, κάνουμε ό,τι μπορούμε για να καταλήξουμε σε ένα καλό σημείο για αυτές τις χώρες. Δεν ανησυχώ ιδιαίτερα, σίγουρα όχι για την Αμίμπεα και για την Κένια τι να πω, να αυτή η επιλογή. Θα σταματήσω εδώ. Είμαι ευγνώμων που υπερασπίζετε το καριφόρομ, αλλά πραγματικά δεν πιστεύω ότι διαιρούμε τις περιφέρειες. Αν ταξιδέψετε στην Αφρική, θα αντιληφθείτε ότι συζητούν διαπεριφερειακό εμπόριο και με άλλους τρόπους και οι ΣΟΕΣ ως περιφερειακή διάσταση σίγουρα βοηθούν να σας δώσω ένα στοιχείο που πραγμα... αποτελεί πραγματική κινητήριο δύναμη είναι το κοινό εξωτερικό δασμολόγιο, το οποίο χρειάζεται ΣΟΕΣ για να μπορέσει να υλοποιηθεί. Μιλήστε στους επιτρόπους της ΕΚΟΒΑΣ, θα σας πούν πόσο επενούν τη διαδικασία ΣΟΕΣ, γιατί αυτή τους συνένωσε ως περιφέρεια. Το ίδιο συμβαίνει και αλλού. Ίσως λιγότερο στην κοινότητα Ανατολικής Αφρικής, γιατί είναι ήδη μια ισχυρή περιφέρεια. Προχωρούν προς μια ενιαία αγορά χωρίς τη βοήθειά μας. Μπορούμε δηλαδή εμεί να εισάγουμε κινητήριε δυνάμει, αλλά δεν μπορούμε να επιθυμούμε αυτές τι κινητήριε δυνάμεις να είναι ισχυρότερε από ό,τι επιθυμούν οι άνθρωποι εκεί. Δεν θα συμφωνούσα λοιπόν με αυτό το ζήτημα του διαχωρισμού, της διαίρεσης. Ε, τέλος, αν και φεύγει τώρα ο κύριος Στέρτη ε, για την Γεωργία. Ναι, παρατηρείται κινητικότητα στη Γεωργία και εμείς ε, ναι, προχωράμε, βρισκόμαστε σε πολύ καλό σημείο και ελπίζουμε ότι θα ολοκληρώσουμε αυτό το κεφάλαιο για τα καλά ε, πολύ σύντομα. Ε, Ευχαριστούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για όλες αυτές τις εξηγήσεις και την ενημέρωση για την κατάσταση. Οι φίλοι της Πολιτικής Ένωσης το παρακολουθούν στενά. Εδώ κλείνει το δημόσιο κομμάτι της ε, συνεδρίασής μας. Το επόμενο σημείο θα ε, διεξαχθεί και κλεισμένο των θυρών. Να ζητήσω λοιπόν σε όσους δεν έχουν το δικαίωμα να παραμείνουν να εγκαταλείψουν την αίθουσα. Ε, next meeting will be in... Η επόμενη συνεδρία θα λάβει χώρα 1η Απριλίου 2014. Θα είναι η τελευταία μας συνεδρίαση πριν από τις εκλογές.